είπα της εκπροσώπου για την ε, διάσκεψη αναθεώρησης του 15 της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η κυρία Μογκερίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή. Αποδίδω μεγάλη σημασία στην διάσκεψη της ε, συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών οπλών που θα γίνει στη Νέα Υόρκη από 22 Απριλίου μέχρι 22 Μαΐου που είναι το σημαντικότερο γεγονός για τον αφοπλισμό φέτος και είχα πει στη σχετική ακρόαση του Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο ήδη πως σκόπευα να εργαστώ πάρα πολύ σκληρά σε αυτό το θέμα και θα πάω στην ε, αρχική διάσκεψη και θα απευθυνθώ στην συνέλευση. Επίσης, θεωρώ πως είχε παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Το 2010 είχε εγκρίνει ένα ψήφισμα που βοήθησε να συνδιαμορφώσει την ευρωπαϊκή θέση και νομίζω πως ε, καλό θα είναι να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος έτσι ώστε η θέση μας να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή θέση και θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω και για όλες τις ε, ε, φορές ε, στις οποίες, τις οποίες προσκαλέσατε την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στην σχετική επιτροπή. Τώρα, για την διάσκεψη αυτή αναθεώρησης της συνθήκης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το επίπεδο εφαρμογής του σχεδίου δράσης του 2010 απόψεις οι οποίες είναι δύσκολο να συμβιβαστούν και θα πρέπει ακριβώς να μην ε, ξεχνάμε κάποια ζητήματα που είναι περιφερειακά και θα ε, έχουν σημασία για τη διάσκεψη αφενός οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν την οποία διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ προσωπικά μετά από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα μπορούσε να αποδείξει πως είναι δυνατή μια ειρηνική λύση η οποία θα είναι αμοιβαία υποφελής και ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της διάσκεψης είναι πως η διάσκεψη για τα όπλα μαζικής καταστροφής ε, και την μη διάδοσή του στην Μέση Ανατολή που ήταν ένα βασικό κομμάτι του σχεδίου δράσης του 2010 δεν έχει ακόμα λάβει χώρα και να σας ευχαριστήσω εδώ πέρα για τις προσπάθειές σας και ελπίζω τελικά να συγκληθεί μια διάσκεψη νωρίς. Όσον αφορά τώρα το σκέλος του αφοπλισμού, υπάρχει μια συζήτηση που λαμβάνει η χώρα κυρίως εκτός των συναντήσεων για το θέμα των καταστροφικών συνεπειών οποιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων και μια μεγάλη συζήτηση έγινε πρόσφατα στην Βιέννη, ε, την οργάνωσε η Αυστρία και κάποιοι βεβαίως θέλουν να μιλήσουν για μια νομική απαγόρευση αλλά άλλοι θέλουν να πάνε σε μια σταδιακή προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον ασφαλείας. Είναι μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται και ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφορετικά κρατημένα με διαφορετικές ιστορίες και ευαισθησίες ε, θα έλεγα. Με ενθάρρυνε πρώτα απ' όλα το ότι κατά την πρόσφατη διάσκεψη στο Λονδίνο τα πέντε κράτη-μέλη της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά και συνεισέφεραν περαιτέρω στην οικοδόμηση της αμοιβιάς εμπιστοσύνης και διαφάνειας ε, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τον πολυμερή αφοπλισμό θεωρώ πως η ε, διάσκεψη, παρά το ότι όπως είπα ακόμα διαμορφώνουμε τη θέση μας, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει ένα όρομα για το πώς θα ενισχύσουμε την συνθήκη συνολικά. Προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη την κοινή μας θέση για τη διάσκεψη και θεωρώ πως ακόμα και αν τα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικά, δηλαδή υπάρχουν κράτη-μέλη με πυρηνικά, μέλη του ΝΑΤΟ, ουδέτερε χώρες κτλ. Είμαι αισιόδοξη πώ θα καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Προσωπικά θεωρώ, αλλά αυτή είναι και η θέση τη ένωση. πως η συνθήκη αυτή είναι και πρέπει να παραμείνει σε μέλος λήθος του Παγκοσμίου Καθιστώτος Μη Διάδοσης. Και του πυρηνικού αφοπλισμού και είναι επίσης σημαντικό στοιχείο στην ε, περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Όπως ξέρετε, εμείς στηρίζουμε την ε, παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή της συνθήκης αυτής και θεωρώ πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε μια πιο συνολική και ισορροπημένη και διαρκή εφαρμογή του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε το 2010 στην διάσκεψη το σχέδιο δράση το οποίο αποτελεί τον κοινό μας οδικό χάρτη εν ώψη της ε, διάσκεψης της Νέας Υόρκης. παρόλα αυτά θεωρώ πως θα καλέσουμε ε, όλα τα συμβαλόμενα μέρη να ανταποκριθούν στις, στις ε, δεσμεύσεις του 2010 και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό όρομα για το πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι δεσμεύσεις. Τώρα γνωρίζω πως δεν έχουμε τόσο χρόνο, αλλά θα ήθελα να περάσω σε κάποιες λεπτομέρειες της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τους τρεις πυλώνες. Πάντα υπό την αίρεση ότι η θέση αυτή ακόμα δεν είναι ε, επίσημη. Για τον αφοπλισμό. Πρέπει νομίζω να επαναβεβαιώσουμε πως είναι δέσμευσή μας να προωθήσουμε τον πυρηνικό αφοπλισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της ε, συνθήκης ε, και να επιτύχουμε συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά την μείωση, την συνολική του παγκοσμίου αποθέματος πυρηνικών Αυτό ιδιαίτερα αφορά την ευθύνη των κρατών μελών που έχουν τα μεγαλύτερα οπλοστάσια και βεβαίως ε, καλωσορίζουμε τις ενδείξεις προόδου από ΙΠΑ και Ρωσία για μια νέα συνθήκη START και του ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν σε περαιτέρω μειώσει του πυρηνικού οπλοστασίου του. Ε, και αυτό αφορά στρατηγικά και μη όπλα, ανεπτυγμένα ε, και μη. Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε επίσης ε, τις διασκέψεις των πυρηνικών κρατών, μεταξύ των οποίων και τις δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διαφάνειας και πιστοποίησης και θα παραμείνουμε δεσμευμένοι στην ανάγκη ελέγχου των όπλων και ενίσχυση των πολυμερών προσπαθειών σε διαπραγματευτικούς φορείς, ειδικά όσον αφορά την διάσκεψη για τον αφοπλισμό καθώς ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ένα πρόγραμμα εργασίας, κάτι το οποίο είναι οπωσδήποτε απαράδεκτο. Και θεωρώ πως θα πρέπει να ζητήσουμε την άμεση έναρξη και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην διάσκεψη του αφοπλισμού για την συνθήκη η οποία απαγορεύει την παραγωγή σχάσιμου υλικού για πυρηνικά όπλα ή άλλες τέτοιες ε, συσκευές και διατάξεις. Κάτι άλλο στο οποίο είμαι προσωπικά ενεργή είναι η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών που είναι βεβαίω πάρα για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό και θα συνεχίσω προσωπικά να εργάζομαι για να τεθεί ενισχύ προφανώς ε, όχι μόνο μου αλλά εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω θα πρέπει να δούμε όχι μόνο την διπλωματική δράση αλλά και την ε, οικονομική δράση και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξη και την χρηματοδότηση που δίνει στην ΚΕΠΑ. Όπως είπα, προσωπικά εγώ εμπλέκομαι στις προσπάθειες που κάνει ο σχετικός οργανισμός σε σχέση με τα κράτη του παραρτήματος 2, τον οποίων η υπογραφή απαιτείται για να τεθεί η συνθήκη ενισχύ. Όσον αφορά τη μη διάδοση, κατά την άποψή μας η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στο μέτωπο της διάδεσης. Είναι πρόφανες αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ακριβώς για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα και ε, ο κύρος της συνθήκης. Τώρα δεν θα αναφέρω συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, μη συμμόρφωσης φαντάζομαι θα τα θίξετε στις ε, παρεμβάσεις σας. Όσον αφορά τώρα την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναβεβαιώσει την στήριξή της για το δικαίωμα όλων των συμβαλωμένων μερών να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια για ε, ειρηνικούς σκοπούς χωρίς καμία διάκριση όσον αφορά την ε, συνθήκη. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό θα ήθελα να αναφέρω την πυρηνική ασφάλεια η συνθήκη κορυφής για την πυρηνική ασφαλεία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ προσωπικά την παρακολουθούσα όταν ήμουν και βουλευτής και υπουργό μετά. Νομίζω πως ε, έχει μεγάλη σημασία για να μειωθεί η απειλή της πυρηνικής τρομοκρατίας, ε, κάτι το οποίο εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία και βεβαίως να εξασφαλίσουμε όλο το ευπαθές πυρηνικό υλικό τα επόμενα χρόνια και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τον ρόλο που παίζει η Διεθνής Υπηρεσία Πυρηνικής Ενέργειας και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα ταμεία πυρηνικής ενέργειας ε, στο οποίο έχουμε συνεισφύρει 40 εκατομμύρια ευρώ από το 2004 και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να σας ζητήσω να συνεχίσετε να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας... Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη. Ανοίγει συζήτηση. Πρώτα θα λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο από το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και είπατε εκπρόσωπε σας ευχαριστώ για την δήλωσή σας και θεωρώ πως το θέμα αυτό υπάρχει ευρύτατη συνένεση εντός της ΕΦΣΑΣ Θεωρώ πως η διάσκεψη αυτή ε, πρέπει να μας βρει ενωμένους ως Ευρωπαίους, πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση. Ελπίζω λοιπόν πως στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Υποστηρίζουμε από βάθος καρδίας τις προσπάθειες των τριών συντριών και θεωρώ πως θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την χώρα αυτή ε, που θα έχει συνολική επίδραση στην διαδικασία της μη διάδοσης. Ανησυχώ τώρα εγώ για μια άλλη χώρα, τη Βόρεια Κορέα και τις πυρηνικές δοκιμές. Δεν τηρεί την απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών, είναι μια χώρα απρόβλεπτη και θα πρέπει να παραμείνουμε σε στενή επαφή με την Κίνα η οποία ε, από ό,τι φαίνεται μπορεί να συγκρατήσει την Pyongyang. Φοβάμαι πως ε, είχαμε ένα πάρα πολύ άσχημο παράδειγμα σε σχέση με την Ρωσία και την Ουκρανία και τα κίνητρα που δίναμε γιατί η συμφωνία της Βουδαπέστης του 1994 είχε όσο βασικό ε, περιεχόμενο ότι θα δώσει τα πυρηνικά της η Ουκρανία και θα εγγυηθούν τα σύνορά της ε, οι μεγάλες δυνάμεις ΙΠΑ ε, και Βρετανία. Και βεβαίως ε, βλέπετε πως αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αντικίνητρο για να παρατήσουν κάποιες χώρες τα πυρηνικά όπλα. Το βλέπουν και σκέφτονται πως θα ήταν καλύτερο να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Δεν είναι λοιπόν αυτό προς το συμφέρον μας και Άρα θα πρέπει να επιστρέψει η Ρωσία στο δρόμο της ειρήνης στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Αναγκόμες, παρακαλώ. 70 χρόνια μετά το ε, γεγονός ότι φτάσαμε σε μία ημερομηνία ρώσιμο για τη Χειροσύμα και Ναγκασάκη βλέπουμε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να αρθεί η χρήση των πυρηνικών όπλων και όχι μόνο στα πλαίσια της αναθεώρησης. Ε, ζούμε μία εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία που προκάλεσε μία πυρηνική δύναμη. Ρωσία με βάση το πρωτόκολλο της Βουδαπέστης του 1984. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική μιλάμε για ένα μεγάλο πόλεμο για την απόκτηση των πυρηνικών όπλων. Δεν είναι αποτρεπτικά τα πυρηνικά όπλα. Η διάδοση οδηγεί σε ολοένα μεγαλύτερη διάδοση, γι' αυτό θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και τη στάση του Ισραήλ, της Βόρειας Κορέας και ούτω καθεξής. Δυστυχώς η Ρωσία, η Κίνα, η ΙΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι παλαιές χώρες κατά κάποιο τρόπο, απέτυχαν αλλά και οι νεότερες αυτές δηλαδή που απέκτησαν τα πυρηνικά όπλα αργότερα. Θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει και στην περίπτωση της ε, Ινδίας, του Ισραήλ και του Πακιστάν θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ότι θα πρέπει τα συμβαλόμενα μέρη να δεχτούν τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων μέσα στα πλαίσια συνομιλιών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, διπλωματικές μας δυνατότητες έτσι ώστε η μη διάδοση πυρηνικών όπλων να αποτελέσει ένα πραγματικό όπλο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταποκριθούν και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Τζαμπάσκι από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι εντυπωσιάστηκα ιδιαιτέρως από την ζωτικότητά σας από το ότι είστε εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας τόση πολλή ώρα για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Τώρα, η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι η μόνη συνθήκη η οποία εστιάζει τον ενδιαφέρον της στην πρόληψη έτσι ώστε να μην εξαπλωθούν τα πυρηνικά όπλα. Πρέπει να δούμε όμως τι γίνεται και με τον Ισλαμικό εξτρεμισμό, το Ισλαμικό κράτος και την απειλή τελικά όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί να καταλήξουν σε λάθος χέρια. Και η διάσκεψη αναθεώρησης σε αυτά θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή, σας, την προσοχή της ε, τέτοιου είδους όπλα είναι σημαντικά για την εθνική ασφάλεια και την ειρήνη, τη σταθερότητα σε διάφορες χώρες και θα πρέπει να μεριμνήσουμε, να μεριμνήσουμε για την ασφάλεια ε, των χώρων όπου αποθηκεύονται. Βήμα προς βήμα πρέπει να είναι η προσέγγιση και θα πρέπει να συνεχίσουμε την προώθηση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής τεχνολογίας, γιατί αυτή είναι η πιο ε, καθαρή ε, τεχνολογία. Και έχουμε το παράδειγμα του Κοσλοντούι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Λέζινγκ. Να ρωτιέμαι γιατί γίνεται μόνο συζήτηση για αυτό το θέμα και όχι ψήφισμα για ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας. Αυτό θα ήταν το σωστό μήνυμα. Η συνθήκη απαγόρευση των πυρηνικών όπλων ε, ήταν η συνέπεια του βομβαρδισμού της Χειροσύμας και του Ναγκασάκη. απειλή με τα πυρηνικά δεν είναι πολιτικό ή στρατιωτικό μέσο και δεν επιτρέπεται να γίνει ποτέ ξανά. 20 χρόνια όμως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου η γη ε, εξακολουθεί να έχει χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο αυτή τη συνθήκη. Αντιθέτως πρέπει να συζητήσουμε τι ρόλο μπορεί να παίξει και θέλει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οπωσδήποτε αδιαμφισβήτητο πως υπάρχουν σκληροπυρηνική σε διάφορες πλευρές. Και το είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες ε, από η Παρουσία, Μεγάλη Βρετανία και Κίνα, οι οποίες έκαναν μια κοινή δήλωση υπέρ του αφοπλισμού. Όμως φαίνεται πως ε, δεν ενδιαφέρει, ε, δεν αφήνει μόνο εμάς αδιαφορούς, αλλά και τον τύπο. Δεν αναφέρεται στον τύπο. Ενώ ακριβώς αυτή την εποχή μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και να ενισχύσει την θέληση για ειρήνη. Αυτό το οποίο χρειάζεται ο κόσμος μας είναι ενίσχυση της λογικής και μια πολιτική ύφεση. Γιατί τα ατομικά όπλα τελικά μας απειλούν όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί είπατε εκπρόσωπε, γνωρίζω ότι υπάρχει μια κοινή θέση και από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Πίτροπε, θα θέλατε να συνεργαστούμε ευρέως και να φτάσουμε και σε ένα κοινό ψήφισμα. Φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο όμως δεν θα φτάσει σε ένα κοινό ψήφισμα. Άρα απομακρυνόμαστε από τη στάση του παρελθόντος. Θα ήθελα να υποστηρίξετε όμως συνάδελφοι μία κοινή πρόταση ψηφίσματος. Όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ, συμφωνούμε σε αδρές γραμμές. Γιατί να μην υποστηρίξουμε την Επίτροπο, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Από τη δική μας πλευρά η συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να αποδυναμωθεί. Οργανώσαμε μία κρόαση στην ε, Επιτροπή μας. Ε, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και φαίνεται ότι οι εταίροι που συμμετέχουν στην ε, συνθήκη το 2015 ίσως δεν θα δεχτούν το πρόγραμμα δράσης που ε, εγκρίθηκε το 2010. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη, δεν νομίζω ότι θέλουν ε, να απορρίψουν συμφωνία, αλλά βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Η κατάσταση έχει αλλάξει ε, προς δυσμάς και στο νότο και δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. Γι' αυτό δεν θα, υπάρξει, δεν θα πρέπει να υπάρξει αναρχία σε έναν μη ελεγχόμενο κόσμο. Κύριε Μογκερίνη, θα ήθελα να κάνετε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε να έχουμε σωστή προσέγγιση στη διάσκεψη, να είμαστε ένα σημαντικό εμπλεκόμενο μέρος και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την συνθήκη αυτή. Από το FTD, ούκεμ, ούκεμ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Από την υπογραφή της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, πολλή δουλειά έχουν κάνει υπογράφοντες για να καταργήσουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν μας ανακούφισε από την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου και πάντοτε υπάρχει κίνδυνος να διαδοθούν και σε περισσότερες χώρες και σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό κάνει την κατάσταση χειρότερη. Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν πόσο γρήγορα μπορεί να καταρρεύσει η ασφάλεια. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι θέμα ασφάλειας και άμυνας ενός κράτους μέλος. Είναι πολύ σημαντικό για την εθνική βρετανική ασφάλεια το επίπεδο του πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης να παραμείνει ε, στα ε, χέρια η απόφαση γι' αυτό ε, του κράτους μέλους και όχι άλλων. Ο κύριος Φρουντζούλικα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω τα θετικά δεν υπάρχει πρόοδος και αυτό δείχνει ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι στη διάσκεψη αναθεώρησης των συμβαλόμενων μερών στη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, ένα θετικό στοιχείο μας δίνει την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Ε, ε πρόοδος υπάρχει στις συνομιλίες με το Ιράν από την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Οι βασικές διαφωνίες φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με ένα κοινό ε, περιεκτικό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και να έχουμε δικλείδης ασφαλείας. Μια τέτοια Ισφανία, συμφωνία μπορεί να γίνει διεθνής κανόνας και ε, να ενθαρρύνει τις συνομιλίες. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια από πλευράς ε, πυρηνικών κρατών. Όλα αυτά είναι θεμελιώδη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτά είναι λοιπόν τα καλά. Ας μιλήσουμε τώρα για τα κακά το Memorandum, το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, το οποίο έχουμε αναφέρει και είναι του 1994, οδήγησε τελικά στο γεγονός η Ουκρανία να παραιτηθεί των πυρηνικών σε αντάλλαγμα ε, εγγυήσεις για την ασφάλεια και αυτό θα υπονομεύσει την ε, διαδικασία για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η κατάσταση στην Ουκρανία δηλαδή όσο κλιμακώνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την υπομονή και τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ ο κύριος Γιούρεκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα πρέπει να καταπολεμήσουμε την διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε ε, και τη δράση των χωρών που απειλούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, γιατί πολύ συχνά αυτά είναι εργαλεία σε αυτή την πολιτική του τρόμου για παράδειγμα, η Ρωσία έχει στρατιωτικό δόγμα και λέει ότι δίνεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα έναντι άλλων ε, κρατών σε περίπτωση πολέμου. Επομένως, είπα ότι εκπρόσωπος της εξωτερικής ε, πολιτικής, περιμένω από εσά να ασκήσετε σφοδρή κριτική σε αυτή την άποψη, διότι η ρωσική θέση αποτελεί απειλή και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρξει σαφής δήλωση ότι μια χώρα σαν τη Ρωσία δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον ενό κράτου που δεν διαθέτει πυρηνικά. Αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Σα ενθαρρύνω να το πράξετε και καλό την Ευρώπη να υιοθετήσει μια τέτοια πρωτοβουλία στην επόμενη διάσκεψη. Ο κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλάμε για συνθήκη για μη διάδοση πυρηνικών όπλων και μιλάμε για ακρόνημα τα οποία ε, δεν γνωρίζει ο μέσος πολίτης όταν μιλάμε για αυτές τις ε, συμφωνίες οι οποίες είναι ύψης της σημασίας. Και εδώ αναφέρομαι στους πέντε στο Συμβούλιο Ασφάλειας που έχουν δικαίωμα βέτο, για να μην μιλήσω για την ε, Βόρειο Κορέα, την, ε, το Πακιστάν και την Ινδία. Μιλάμε για θέσεις που δεν δικαιολογούνται πάντα στο, στο Όσλο και στη Βιέννη το είδαμε αυτό. Θα πρέπει να ζητήσουμε την απομάκρυση των πυρηνικών όπλων που θα πρέπει να είναι κοινό μας μέλημα και για όλους όσους κατέχουν τέτοια οπλοστάσια. Ξέρουμε ποιο είναι το γεωπολιτικό παιχνίδι της Ουκρανίας. Θα πρέπει να έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο και πιστεύω ότι ως προς το CTBT θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά Μάρσαλ. Ας ρωτήσουμε τους κατοίκους κατά πόσο χρειάζεται να σταματήσουν οι δοκιμές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και μία αποζημίωση, να δοθεί αποζημίωση από τις ΗΠΑ. Κούφοντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Αντιπρόεδρε για την δήλωση που κάνατε για τη μη διάδοση Πλέον δεν είναι πρωτοσέλιδη η είδηση αυτό το θέμα. Στη γενιά μου και σε κάποιους άλλους ε, μοιάζει ένα πρόβλημα του παρελθόντος και του ψυχρού πολέμου. Όμως ε, τώρα οι εντάσεις μεταξύ των πυρηνικών κρατών έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες. Ε, γίνεται ένας πόλεμος διατυπωσόπου με την Ρωσία, Ανατολή και Δύση και πάλι ε, βρίσκονται σε σύγκρουση και οι Αμερικανοί συμμαχοί μας σκέφτονται να στείλουν όπλα και η Ευρώπη ανησυχεί για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και τη μη διάδοση των πυρηνικών. Οι εντάσεις ζητούν και απαιτούν ε, ανανεωμένη εμπιστοσύνη και ίσω και νέε επιθεωρήσεις για την τήρηση των συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το πλαίσιο τη μη διάδοση να μην καταλήξει απλά άλλο ένα φόρουμ για σύγκρουση. Οπότε σα ζητώ να δηλώσετε ξεκάθαρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωση πω οι εντάσει με τη Ρωσία δεν πρέπει να σταματήσουν να επιβραδύνουν ή να εμποδίσουν τα ήδη συμφωνηθέντα όσον αφορά την μείωση των πυρηνικών όπλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπαλτσίτης για ένα λεπτό. sudėtingas Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα των πυρηνικών όπλων είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Και σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη για την αναθεώρηση της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, είναι σαφέστατο ότι μια εύκολη λύση δεν θα ε, υπάρξει. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί λύση. Αυτό σίγουρα ισχύει. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα κάνει η, Βόρεια Κορέα, Βόρειος Κορέα, για παράδειγμα. Σήμερα μπαίνουμε τώρα σε ένα άλλο στάδιο και θα ήθελα να αναφερθώ στην κρίση στην Ουκρανία και στη θέση της Ρωσίας. Η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων ε, διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπου υπήρχε σταθερότητα τρόπον τεινά. Ε, σε κάθε περίπτωση, σήμερα οι προσπάθειες μας υπέρ της σταθερότητας ας ελπίσουμε ότι θα είναι καρποφόρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπενιφέη, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη φορά δεν θα παρουσιάσουμε, δεν θα υποβάλουμε κοινή πρόταση ψηφίσματος ε, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν γινόταν κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα την περίοδο 2005-2010. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε και σε μια συμφωνία με το Ιράν για τη χρήση πυρηνικών όπλων πέρα από την κατάσταση, την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία. Δεν ε, μιλάμε για μια μακροχρόνια συζήτηση. Πιστεύουμε ότι η μη διάδοση έχει μεγάλο αντίκτυπο στην εξωτερική μας πολιτική, γι' αυτό και χάσαμε μια ευκαιρία. Αυτό όμως δεν ε, σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεύρουμε νέους δρόμους και δεν πρέπει να ξεχνάμε τη διάσκεψη της Βιέννης, η οποία έδωσε μια νέα όθηση ε, για 44 χώρες. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τη μη διάδοση μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Στα πλαίσια του Catch the Eye World για ένα λεπτό. Νέα φακολτά. Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο. I νόμιζα ότι είπατε κύριος Ward, εγώ είμαι η κυρία Ward. Συνεργάζομαι στενά με την κοινωνία των πολιτών, η οποία ανησυχεί ιδιαίτερα ε, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και οι χώρες που δεν έχουν πυρηνικά όπλα ανησυχούν ιδιαίτερα για την απειλή που αποτελούν τα πυρηνικά όπλα. Μαζί με πολιτικούς εκπροσώπου από πάνω από 160 χώρε πήγα στην διάσκεψη της ε, Βιέννης ε, που διοργάνωσε η Αυστριακή Κυβέρνηση για να δούμε ακριβώς ε, τις συνέπειες των πυρηνικών όπλων και βεβαίως πριν από αυτό είχαμε και το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών. Οι οργανώσεις αυτές και οι άνθρωποι που εκπροσωπούν πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για τη μη διάδοση και την πιθανή απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Σας ευχαριστώ γιατί τηρήσατε και το χρόνο σας. Γιακοβίτς, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι είπαν ότι χρειαζόμαστε ένα ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ εδώ πέρα πως πρέπει να είναι ενωμένο να αντιληφθούμε τον κίνδυνο των πυρηνικών όπλων όχι μόνο γιατί μπορούν κάποιες χώρες να τα χρησιμοποιήσουν κατά της δημοκρατίας ε, και όλων των αρχών μας αλλά γιατί πλέον ε, με τα πυρηνικά όπλα αμφισβητείται ολόκληρος ο κόσμος Ακούγοντας λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ανέφερε η κυρία Μογκερίνη, δηλαδή μικρότερα από θέματα πυρηνικών κεφαλών, περισσότερη ασφάλεια, πρέπει τουλάχιστον να έχουμε ένα νομίζω, πρόγραμμα, ε, νομίζω πράγμα την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ο αφοπλισμός είναι ύψης της σημασίας γιατί θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, Συμφωνία Μη Διάδοσης ε, Πυρηνικών Όπλων. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι διεθνώς. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε και το γράμμα και το πνεύμα της συνθήκης. Θα πρέπει λοιπόν να μην δεχτούμε τη χρήση αυτών των ε, οπλοστασίων η ΕΠΑ και το ΝΑΤΟ ε, θα πρέπει να απαρνηθούν τη χρήση αυτής της δύναμης. Και αυτό αφορά και την Ευρώπη και την Ασία. Πιστεύω ότι η είπα προώθησαν μία νέα πολιτική, την πολιτική Ομπάμα, ε, του Ομπάμα, ο οποίος όμως χρησιμοποιεί μία ε, γλώσσα υποκρισίας. Δείτε τι συνέβη στο Ισραήλ, το οποίο δεν προσυπέγραψε τη συνθήκη και ε, ζει σε κατάσταση ατιμορρησίας σε αντίθεση με το Ιράν. Είναι πολύ λυπηρό διότι οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες, το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές δεν ήθελαν να εγκρίνουν μια πρόταση ψηφίσματος για τη συνθήκη αυτή. Λίγη τώρα η συζήτηση, το ο κύριος Κοράου ζήτησε το λόγο και εκείνο ε, για ένα λεπτό και είναι και η τελευταία παρέμβαση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι με, ότι με ξεχάσατε. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μία συνθήκη και την αναθεώρηση της συνθήκης μη διάδοσης πυρηνικών όπλων που θα γίνει το Μάιο του 2015 και είναι λυπηρό για το, ότι μιλάμε για πυρηνικά όπλα 70 χρόνια μετά το Ναγκασάκι και τη Χειροσύμα. Πολλές ε, μη ε, δυτικές χώρες στην ουσία επιδίδονται σε έναν αγώνα απόκτησης πυρηνικών όπλων. Γίνεται λόγος για εγγύηση της ασφάλειας μέσω των πυρηνικών, μα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τα πυρηνικά θα πρέπει να εξαφανιστούν από προσώπου γης. Εμείς διπλωματικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καμία δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν και η τελευταία παρέμβαση. Το λόγο έχει η Αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μογκερίνη. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με μία παρατηρήση από τις τελευταίες παρεμβάσεις που ήταν σαφέστατη και τα είπε όλα. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη συνθήκη, να την ενισχύσουμε και να διασφαλίσουμε ότι θα ε, γίνουν όλες οι χώρες μέλη σε αυτή θα προσχωρήσουν σε αυτήν και θα την εφαρμόζουν και στην ουσία και επί των τύπων. Αυτό είναι ο πυρήνας του ευρωπαϊκού μηνύματος. Αυτό θα διαλαλήσουμε στη διάσκεψη για την αναθεώρησή της. Και είπατε επίσης, ε, αναφερθήκατε σε διαφορετικές γενιές και στο παρόν και στο παρελθόν και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό φαίνεται προφανές και ακούγεται προφανές σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους ότι δεν θα πρέπει καν να συζητείτε αυτό το θέμα, ότι είναι τόσο προφανές που δεν χρειάζεται καν να συζητηθεί. Ωστόσο, ε, πρέπει να διανύσουμε ακόμα αρκετή απόσταση για να φτάσουμε εκεί. Σίγουρα πολλά μένουν να γίνουν στον πυλώνα της μη διάδοσης των πυρηνικών οι διαπραγματεύσεις για το, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σίγουρα θα έχουν αντίκτυπο στη διάσκεψη αυτή καθεαυτή. Ελπίζω ότι θα έχουν υπάρξει αρκετές θετικές εξελίξεις μέχρι τότε και σας διαβεβαιώ ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί και κάνω ε, Δίνω τον καλύτερο εαυτό μου για να υπάρχει θετική έκβαση στις συνομιλίες. Είναι μια ιστορική ευκαιρία αυτή, γιατί έχουμε μιλήσει για τον αφοπλισμό, αλλά ο πυλώνας για τη μη διάδοση είναι εξίσου σημαντικός με τον αφοπλισμό. Και μάλιστα νομίζω ότι ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και έτσι μπαίνουμε σε ένα ενάρετο κύκλο αξιοπιστίας. Και γι' αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Να αναφέρω δύο πράγματα που σίγουρα μένουν από αυτή τη συζήτηση. Το θέμα του ψηφίσματος σας αφορά αποκλειστικά και μόνο εσάς, όχι εμάς. Ωστόσο, θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι ενθαρρυντική, θέλετε να με ενθαρρύνετε και σας ευχαριστώ και θέλω να διατηρηθεί πραγματικά αυτή ο διάβλος επικοινωνίας διαμέσου των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πρώτον, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα έχει ε, μία πολύ σημαντική ε, φωνή που πρέπει να ακούγεται και δεύτερον διότι είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν την ε, κοινωνία των πολιτών, με την κοινή γνώμη και με τα εθνικά κοινοβούλια μέσω ημών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη δική σας δουλειά μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι σημαντικό γιατί είναι ένα θέμα που επηρεάζει ιδιαίτερως την ασφάλεια των πολιτών. Ξέρετε, πολύ συχνά υπάρχει ψευδέστηση ότι η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων έχει να κάνει με την καλή βούληση ή τα τα πολύ θετικά συναισθήματα και την καλή διάθεση ορισμένων αφελών ή πολλών αφελών αν θέλετε. Ενώ ε, την πραγματικότητα αυτή η συνθήκη έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια. Ακριβώς λόγω των ε, απειλών και της έντασης που υπάρχει σε θέματα ασφαλείας, στοιχεία τα οποία όλο και οξύνονται και όλο και εντείνονται, ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε να ε, δουλεύουμε πάνω στην εφαρμογή της συνθήκης, να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα, να δώσουμε συνέχεια στα ε, ε, βήματα που έχουν γίνει τις περασμένες δεκαετίες και ούτω καθεξής. αναφερθήκατε στην, στο δόγμα του Ομπάμα και στην ομιλία της Πράγας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά Ξέρετε, οι εντάσεις που υπάρχουν, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού, ε, τραβούν την προσοχή από τον πραγματικό ε, σκοπό της δουλειάς μας για τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και των συνοδών ε, συνθήκων. Πραγματικός μας σκοπός και στόχος και τη συνθήκη άλλωστε είναι να αυξήσουμε την ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι να τη μειώσουμε θα κάνουμε το παν έτσι ώστε να μιλήσει η Ευρώπη με μία φωνή και μάλιστα χειρή στη διάσκεψη αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία ε, Μογκερίνη. Σας ευχαριστώ για αυτό τον σημερινό μαραθώνιο, σήμερα το απόγευμα. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις, ακούστηκαν και πολλά αρνητικά για ε, εμάς, για το Προεδρείο, κάτι το οποίο θα αποτιμηθεί.